Σα, λοιπόν, αφήστε το παιδί σα. Δεν θα σα πω Δεν θα σα πω ότι είναι κοντά στο παιδί σα. Δεν θα σα πω ότι είναι κοντά στο παιδί svojim revolučným pohybom otvorilo na... Es que todo momento histórico para Europa. Que fueron los primeros que lucharon por la libertad. Ce journal dont les journalistes son tués. This has happened in my own country. Devletin varlığı ve bağımsızlığı 这完全是因为很多的朋友的帮助。Je prends ici la parole qu'on me confisque dans mon pays. Kosovo se trouve dans une situation extrêmement dramatique. του Centro de Poder Democrático. Cargos electos no nacionalistas son asesinados. A sustained dialogue of tolerance. Andrei Saharov al pueblo de Cuba. The situation is all the more tragic. На свободную, нет цензурированную has to be reformed and it has to be reviewed. премия так молодых лидеров. Gives me the opportunity to speak to you. 状态就是说警察围困的状态。В вообще на Северном Кавказе. Cuando vas a permitir las The spectre of war is haunting our world. Still, there is hope. C'est dramatique, il faut que ça s'arrête tenemos que tener libertad. Il presidente et madame Joël Ilham, représentante de monsieur Ilham Toti. Ο πρόεδρος και πρόσωπος του κυρίου Ilham Toti. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Χαίρομαι πολύ που είμαι στη θέση να ε, καλωσορίσω την κόρη του Λιαμ η οποία ήρθε σήμερα εδώ για να εκπροσωπήσει τον πατέρα της σε αυτή την τελετή απονομή του βραβείου Σαχάροφ για την ελευθερία σκέψης για το 2019. Ε, θα ήθελα να απευθυνθώ ε, και να ευχαριστήσω όλους όσοι ήρθαν στην τελική φάση της επιλογής του βραβείου ε, που ε, παρουσιάστηκαν, που προτάθηκαν από τους ευρωβουλευτές μας και είναι σήμερα κοντά μας, βρίσκονται όλοι στο θεωρείο. Έχουμε εκπροσώπους ε, της Βραζιλίας του, του κινήματος για την διατήρηση της φύσης, για την προστασία του Αμαζονίου. Την Μόνικα Μπενίτσο, την εκπροσώπηση της Μαριέλ Φράνκο που δολοφονήθηκε τον Μάρτιο του 2018. Κλοντελίσε Σίλβαντο Σάντος. Πάτσουν Μεκτουντήρε που εκπροσωπεί τον κάπο Ραόνι, τον παππού της. και για τους ε, restorers έχουμε νέες ε, φοιτήτριες ε, οι οποίες, από την Κένια οι οποίες αποφάσισαν να χρησιμοποιήσουν την τεχνολογία για τη χειραφέτηση των γυναικών και για τον αγώνα κατά του ακροτηριασμού των γεννητικών οργάνων των γενών. Στάζι Ουίνο, Σίτσια Οτιένο, Πούριτι Ούμα, Μακρίν Ονιάγκο εκ μέρους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθατε σήμερα κοντά μας και σας συγχαίρουμε για το θάρρος σας και για την απόλυτη δέσμευσή σας και βεβαίως θα συνεχίσουμε να παρακολουθούμε τις δραστηριότητές σας. Πριν λοιπόν προχωρήσουμε, θα ήθελα να σας παρακαλέσω να παρακολουθήσουμε ένα σύντομο βίντεο για τον νικητή της φετινής χρονιάς του βραβείου Ζαχάροφ, τον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 Κυρίες και κύριοι, αγαπητοί συνάδελφοι, ε, σήμερα λοιπόν απονέμουμε το βραβείο Ζαχάροφ για την ελευθερία της σκέψης ε, στον καθηγητή Ιλαμτότη, ο οποίος δυστυχώς δεν μπορεί να είναι σήμερα κοντά μας, διότι κρατείται στη φυλακή από το 2014. Ο αγώνας του, για την οποία καταβάλει ακόμα ένα πολύ ε, ακριβό τίμημα, υψηλό τίμημα, είναι για μας πηγή έμπνευση και εκφράζω τις θερμές μου ευχαριστίες στην κόρη του, την κυρία Τζουερ η οποία είχε το θάρρος να έρθει εδώ για να τον εκπροσωπήσει. Έτσι λοιπόν, στην καρδιά της Ευρωπαϊκής Δημοκρατίας μπορούμε να ακούσουμε και να αισθανθούμε, κυρίως να ακούσουμε βέβαια, τη φωνή εκείνων ε, που δεν μπορούν ε, να εκφραστούν ελεύθερα στις χώρες τους. Με την απονομή του βραβείου Ζαχάροφ, αυτό το κοινοβούλιο γίνεται ε, εκπρόσωπος της ελευθερίας της σκέψης και του λόγου, μια ελευθερία ιδιαίτερα πολύτιμη για πάρα πολλούς ανθρώπους που δυστυχώς ακόμα αντιμετωπίζουν πολλούς κινδύνους. Είμαι λοιπόν ε, ιδιαίτερα χαρούμενος και νιώθω ότι είναι τιμή για μένα το ότι μπορώ να απονείμω το ε, βραβείο αυτό ε, στον καθηγητή Λαμπτότη, ο οποίος αγωνίζεται για το διάλογο, για την κατανόηση, για την πετριοφροσύνη, τη συμφιλίωση, για την πολιτιστική διαφοροποίηση. Είναι ίδιες αξίε οι οποίε βρίσκονται στην βάση του ευρωπαϊκού Εγχειρήματο ο κύριος Τότι είναι καθηγητής οικονομίας, είναι όμως μια φωνή που καλεί όλους μας ε, στην ε, αυτοσυγκράτηση, γιατί ο ίδιος αγωνίζεται για τα δικαιώματα της μειονότητας των Ουιγούρων στην Κίνα, ελπίζοντας ότι θα μπορέσει να βελτιώσει τις συνθήκες διαβίωσής τους. Οι Ουιγούροι είναι πάντα θύματα διώξεων, ε, σωματικών διώξεων, πολιτιστικών, θρησκευτικών, οικονομικών, πολιτικών διώξεων. Από τον Απρίλιο του 2017 πάνω από ένα εκατομμύριο αθώων Ουιγούρων ε, αυθαίρετα κρατούνται σε φυλακές ε, όπου είναι αναγκασμένοι να απεκδηθούν της εθνικής τους ταυτότητας ε, και των πολιτικών τους επεπιθήσεων. Αυτός ο λαός είναι λοιπόν ένας μεγάλος λαός με μια ουσιαστική ταυτότητα, με μια ιστορία πάρα πολλών χιλιάδων ετών έχουν ένα πολιτισμό που πραγματικά αξίζει να διαφυλαχθεί. Ο Ήλαμ Τότι μέσα από τις ε, μιλταριστικές του δραστηριότητες προσπάθησε και κατάφερε να τους δώσει φωνή. Ο ίδιος βέβαια είναι στη φυλακή αλλά η φωνή του σήμερα είναι εδώ μέσα από τη φωνή της χώρης του ε, και πολλών άλλων Ουιγούρων. Πάνω από 20 χρόνια ε, αόκνα αγωνίζεται για να προάγει το διάλογο και την αμοιβαία κατανόηση ανάμεσα στους Ιγούρους και τους άλλους ε, λαούς της Κίνας. Ε, παρ' όλα αυτά καταδικάστηκε σε ισόβια κάθυρξη με την ε, κατηγορία της υποκίνησης αποσχιστικών τάσεων. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο απαιτεί την απελευθέρωσή του χωρίς όρους και χωρίς καθυστέρηση. ο αγώνας του και όλα αυτά τα οποία έχει υποφέρει, όλα αυτά μας υπενθυμίζουν ότι οφείλουμε να αγωνιζόμαστε για την ελευθερία της σκέψης. Είναι ένα θεμελιώδες δικαίωμα το οποίο μερικές φορές ε, για να το αποκτήσει κανείς ε, πληρώνει τίμημα ακόμα και τη ζωή του. Βέβαια πρέπει να επενθυμίσουμε και όλους τους άλλους, εκείνους ε, που έχουν κερδίσει σε άλλες περιπτώσεις βραβείου που και αυτοί βρίσκονται στη φυλακή και διώκονται γιατί περασπίστηκαν τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις θεμελιώδεις ελευθερίες. Και μάλιστα μερικές φορές φυλακίστηκαν απλά και μόνο γιατί κέρδισαν το βραβείο Ζαχάροφ. Και αναφέρομαι στον Νασρίν Σοτουντέ, Ραΐφ Μπαντάουι, οι κυρίες στα Λευκά, διάφορα μέλη της Δημοκρατικής Αντιπολίτευσης της Βενεζουέλας, Ασμά Μαφούτς. Αυτό λοιπόν το Κοινοβούλιο θέτει το αίτημα στον ύπατο εκπρόσωπο να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα, ε, κυρίως σε επαφές που έχει με τα διάφορα κράτη, για να επιτύχει την απελευθέρωση και την πάυση δίωξης ε, των νικητών του βραβείου Ζαχάροφ. Αυτό το αίτημα βέβαια απευθύνεται και στα ίδια τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στις κυβερνήσεις μας, διότι στο πλαίσιο των διμερών τους σχέσεων ε, με ε, κάποιες χώρες θα πρέπει να προσπαθούν να μεταφέρουν τις αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να υπερασπίζονται τα ανθρώπινα δικαιώματα και την ελευθερία. Σήμερα θα έπρεπε να είναι η μέρα χαράς για να εορτάσουμε την ελευθερία της σκέψης. Είναι όμως μια θλιβερή ημέρα γιατί στον κόσμο που ζούμε το να είναι κανείς ελεύθερος να σκέπτεται δεν σημαίνει πάντα ότι είναι πραγματικά ελεύθερος. Έτσι λοιπόν, ελπίζοντας ότι ο Ιλαμ Τότι θα αφαιθεί ελεύθερος και θα έρθει να μας βρει εδώ στο Κοινοβούλιο, απευθύνουμε τις σκέψει μας σε εκείνον, στην οικογένειά του, στους συγγενεί του, σε όλου όσους βρίσκονται στις φυλακές. Η κόρη του, η κυρία Τζουρ Ιλάμ, μας κάνει την τιμή να βρίσκεται εδώ για να τον εκπροσωπήσει και ευθύ αμέσω τη δίνω το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Assalamualaikum. Ειρήνη Μην. Θέλω να ευχαριστήσω το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και όλους όσους κατέστησαν δυνατόν ε, ο πατέρας μου να λάβει το βραβείο Ζαχάροφ για την ελευθερία της σκέψης. Έχετε παρουσιάσει και τονίσει όχι μόνο το έργο του πατέρα μου και τη δίωξη που έχει υποστεί, αλλά ε, φαίνεται στην προσοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του υπόλοιπου κόσμου τα δεινά ε, ενό εκατομμυρίου Ιγούρων και πάνω που καταναγκαστικά κρατούνται σε στρατόπεδα συγκέντρωσης ε, στην περιφέρεια των Ιγούρων. Ρεχμέτε, ευχαριστώ. Είναι τιμή μου να βρίσκομαι σήμερα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για να παραλάβω το βραβείο Ζαχάροφ εκ μέρου του πατέρα μου. Σα ευχαριστώ για την ευκαιρία που μου δίνετε να αφηγηθώ την ιστορία του, γιατί δεν μπορεί να την αφηγηθεί ο ίδιο. Για να είμαι ειλικρινή μαζί σα, δεν ξέρω πού βρίσκεται ο πατέρα μου. Το 2017 ήταν η τελευταία φορά που η οικογένειά μου έμαθε νέα του. Τότε κρατήτω στην φυλακή Ουρούμκη. Δεν έχω δει τον πατέρα μου από τότε που μας χώρισαν στο αεροδρόμιο του Πεκίνου του 2013. Ετοιμαζόμαστε να ταξιδέψουμε στο Πανεπιστήμιο της Ινδιάνα, όπου ο πατέρας μου είχε προσκληθεί ως ακαδημαϊκός. Δυστυχώς ε, δεν κατάφερε ποτέ να μεταβεί στις Ηνωμένες Πολιτείες. Την ημέρα εκείνη μας έβγαλαν από την ε, ουρά του ελέγχου, μου δώσανε την επιλογή να μπω στο αεροπλάνο και να πετάξω στις Ηνωμένες Πολιτείες ή να μείνω με τον πατέρα μου. Ο πατέρας μου επέμεινε να συνεχίσω. Μου είπε, μην κλαις. Μην τους αφήσουμε να πιστεύουν ότι τα κορίτσια των Ιγούρων είναι αδύναμα. Έφυγα και βάσει της ενθαρρυσής του και λόγω της ενθαρρυσής του είμαι σήμερα εδώ στο Στρασβούργο μαζί σας. Αλλά ενώ εγώ συνέχισα το ταξίδι μου, αυτός ε, συνελήφθη, ε, ξυλοκοπήθηκε, ανακρίθηκε και τώρα εκτεί μια ποινή ισόβιας κάθριξης σε μια κρυφή τοποθεσία. Δεν θα μπορέσω ποτέ να ξαναταξιδέψω πίσω στην Κίνα και να συναντήσω ξανά την οικογένειά μου. Είναι δύσκολο ε, να πιστέψει ότι ο άνθρωπο εξακολουθεί να μοιάζει εξωτερικά με τον άνθρωπο που ήξερε ω παιδί, για τον άνθρωπο που με τι πιτζάμε του δούλευε στο ε, γραφείο, στο υπνοδωματιό μου, αφού παραπονέθηκα ότι περνούσε περισσότερο χρόνο στην ιστοσελίδα του παρά μαζί μου. Όταν υπήρχε ένα πρόβλημα, πάντοτε είχε μία λύση να μου προτείνει πίστευε πω όταν υπάρχει πρόβλημα θα πρέπει να το διορθώσει. Ε, Όπω όταν έχει τρυπήσει ένα ρούχο, θα πρέπει να το ράψει έναν επίλυτο πρόβλημα, πίστευε, θα οδηγήσει σε μεγαλύτερο πρόβλημα. Και επομένως έφερνε τον υπολογιστή του στο δωμάτιό μου και δούλευε στο γραφείο μου ενώ εγώ καθόμουν στο κρεβάτι και έκανα τα μαθήματά μου. Έτσι μπορούσαμε να είμαστε μαζί. Μερικές φορές ε, θα ξεχνούσε πόσο, πόσο αργά ήταν και ήταν απορροφημένο στη δουλειά του μέχρι τι 4 το πρωί εγώ κοιμόμουν και ξυπνούσα και άκουγα το κλικ των δαχτύλων του στο πληκτρολόγιο. Τότε ήμουν έφηβη. Και δεν καταλάβαινα πολύ γιατί ο πατέρας μου θα εγκατέλειπε την ε, ε, σταδιοδρομία του ε, και τις επισκέψεις μας στην αγορά ε, για μια ζωή που θα τον οδηγούσε στη φυλακή. Υπήρχε μια εποχή που μπορούσαμε να αγοράσουμε ένα ολόκληρο αρνί ε, και να το μοιραστούμε με όλη τη γειτονιά. Αφού ο πατέρα μου άρχισε να περασπίζει τα δικαιώματα των Ουιγούρων, ε, δεν είχαμε και τόσε πολλέ ε, φορέ κρέα ε, στην οικογένειά μα. Ε, ο πλούτος, ε, η περιουσία του πατέρα μου πήγε στην υποστήριξη της κοινότητας των Ουιγούρων, τα άσταγα παιδιά ή τις μητέρες. Όταν αγόρασε εκείνα σερβερ στις Ηνωμένες Πολιτείες για να εξασφαλίσει την ιστοσελίδα του Ιγκουρμπής, δεν είχαμε πλέον χρήματα για να αγοράσουμε αρνή. Ο πατέρας μου δεν φοβόταν τη φτώχεια, αρκεί να μπορούσε ε, να αφιερώσει τη ζωή του στον αγώνα, στο να προωθήσει τον ειρηνικό διάλογο και την κατανόηση μεταξύ των Κινέζων Χάν και των Ουιγούρων που ζουν στο δυτικό τμήμα της Κίνας. Γι' αυτόν το πρόβλημα ήταν ξεκάθαρο. Καταπατούνταν βασικά δικαιώματα των Ουιγούρων. Το δικαίωμα να πιστεύουμε αυτό που θέλουμε να πιστεύουμε, το δικαίωμα να ε, λατρεύουμε με τον τρόπο που θέλουμε και το δικαίωμα να σκεφτόμαστε αυτά που θέλουμε να σκεφτόμαστε. Γι' αυτόν η λύση ήταν απλή να ξεκινήσει μια συζήτηση με την κινέζικη κυβέρνηση για να υπάρχει συνεργασία με το λαό των Ιγούρων με έναν ειρηνικό μη βίαιο τρόπο. Η κινέζικη κυβέρνηση δεν ενδιαφερόταν στο να μπει σε συζητήσει για να μειώσει τις εντάσεις στην περιοχή των Ιγούρων με έναν ακαδημαϊκό όπως ο πατέρας μου, ένας άνθρωπος που επιζητούσε μία η ειρηνική λύση με τους Κινέζους Χάν, για να μπορούμε να ζούμε αρμονικά. Αντίθετα, το έβαλαν την ετικέτα του αυτονομιστή και τον κλείδωσαν στην απομόνωση επειδή ήθελε να δώσει φωνή στους ανθρώπους που ήθελε να ελέγξει η κινέζικη κυβέρνηση. Σήμερα δεν υπάρχει ελευθερία για τους Ιγούρους στην Κίνα, το ξέρετε. Ούτε στο σχολείο, ούτε στο δημόσιο χώρο, ούτε ακόμη και μέσα στα ίδια τα σπίτια. Ο πατέρας μου, όπως οι περισσότεροι γούροι, ε, βαφτίστηκε βίαιος εξτρεμιστής ε, με νόσους που πρέπει να θεραπευτούν και μυαλά που πρέπει να αλλάξουν. Υπό αυτή την ψεύτικη κατηγορία η κυβέρνηση έχει θέσει πάνω από ένα εκατομμύριο ανθρώπους πιθανότητα σε στρατόπεδα συγκέντρωσης. Οι Ουγγούροι αναγκάζονται να καταλήψουν τη θρησκεία τους, τη γλώσσα τους και τον πολιτισμό τους. Και οι ε, άνθρωποι βασανίζονται και αναγκάζονται σε καταναγκαστική εργασία. Κάποιοι έχουν πεθάνει. Η ιστορία επαναλαμβάνεται και δεν είχαμε καλή κατάληξη στο παρελθόν, ούτε και τώρα θα έχουμε η Κίνα τα έχει βαφτίσει ως κέντρα επενεκπαίδευσης. Συγγνώμη, αλλά δεν το δέχομαι αυτό το όρο, ούτε και εσείς θα έπρεπε. Ο εξτρομισμός είναι το είδος της γλώσσας που χρησιμοποιεί η κινέζικη κυβέρνηση για να αιτιολογήσει το ότι χωρίζει οικογένειες, το ότι ελέγχει και παρακολουθεί κάθε κίνηση των υγόρων εντός και εκτός της Κίνας και βάζει τόσο πολλούς αθώους ανθρώπους σε στρατόπεδα. Ακόμη και στο σπίτι μου στην Ουάσιγκτον συχνά χακάρουν το τηλέφωνο και τον υπολογιστή μου. Με ρωτούν διάφοροι άνθρωποι αν φοβάμαι. Ναι, φοβάμαι. Μερικές φορές ε, ξεκινώ, ε, συγγνώμη, ξυπνώ και με λούζει κρύος υδρότας. Ε, μερικές φορές ανησυχώ ότι αυτά που λέω θα βλάψουν την οικογένειά μου στην Κίνα. Ακόμη και το ότι περιβρίσκομαι εδώ σήμερα με αγχώνει και είμαι σίγουρη ότι και ο πατέρας μου φοβόταν. Αλλά όταν εντόπιζε ένα πρόβλημα, ξεπερνούσε το φόβο του εργαζόμενος προς μια λύση χωρίς να λαμβάνει υπόψη το κόστος. Είμαι εδώ σήμερα γιατί θέλω να υποστηρίξω τον πατέρα μου. Επομένως, ε, ζητώ από εσά που βρίσκετε εδώ σε αυτή την αίθουσα, αλλά και όσου μας ακούνε, βλέπετε ένα πρόβλημα με τον τρόπο που η κινέζικη κυβέρνηση μεταχειρίζεται το λαό των Ιγουρών. Αν βλέπετε ότι υπάρχει πρόβλημα, σας παρακαλώ να εργαστείτε προς μία λύση. Να εργαστείτε από τη, σας, από δική σας θέση επιρροής. Στα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να πω, χρησιμοποιήστε την ομοθεσία σας για να λογοδοτήσει η κινέζικη κυβέρνηση στις επιχειρήσεις, να μην είστε συνένοχοι ε, στις διώξεις ε, του λαού των Ιγούρων. Στους ακαδημαϊκούς συνεχίζετε την έρευνά σας ε, για να συνεχίζουν να αποκαλύπτονται αυτές οι εκτινοδίες της ΜΚΟ. Συνεχίστε την καλή δουλειά και να επιμείνετε. Στους φοιτητές να μορφώσετε τον εαυτό σας και ποτέ να μην σταματήσετε να αναζητάτε την αλήθεια και να αγωνίζεστε για τη δικαιοσύνη. Εδώ δεν μιλάμε για αγώνα κατά της Κίνας, μιλάμε για προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Θέλω να κάνω μια ειδική μνήμα στους φοιτητέ ε, του πατέρα μου, οι οποίοι μπήκαν για χρόνια στη φυλακή επειδή υποστήριξαν αυτό και τα σχέδιά του. Οι γενναίοι αυτοί οι άνθρωποι, όπως και τα αδέλφια μου οι Γουροί, δεν είναι μόνοι τους στα στρατόπεδα οι Καζάκοι, οι Ουσμπέκοι και άλλοι άνθρωποι βρίσκονται στα στρατόπεδα συγκέντρωση απλώ επειδή είναι αυτοί που είναι. Οι δικηγόροι ανθρωπίνων δικαιωμάτων και οι υπερασπιστέ ανθρωπίνων δικαιωμάτων κρατούν τη φυλακή επειδή προστατεύουν τα δικαιώματα άλλων ανθρώπων. Αλλού στην Κίνα, ε, οι Κινέζοι χριστιανοί, οι Θεβετιανοί και οι πολίτε του Χονγκ Κόνγκ συνεχίζουν να αγωνίζονται για να προστατεύσουν την ταυτότητά του και τα ανθρώπινα δικαιώματα υπό το πνεύμα της δουλειάς του πατέρα μου για να προωθήσουμε την κατανόηση και το σεβασμό μεταξύ των διάφορων κοινοτήτων ε, θα ήθελα ε, να απευθυνθώ και στους άλλους ε, φιναλίστ. Πρέπει να δώσουμε προσοχή και στο δικό τους έργο ακόμη και αν δεν έχουν λάβει το βραβείο. Σας ζητώ λοιπόν να καλύψουμε περισσότερο για τους ριστόρερ που κάνουν εξαιρετική δουλειά για να βελτιώσουν τη ζωή των γυναικών στην Κένια και αλλού στην Αφρική, στη Βραζιλία, τον αγώνα της ε, Μαριέλ ε, Φράνκο, του αρχηγού Ραονί και της κυρίας Σίλβαντο Σάντος. Οι αγώνες τους θα πρέπει να υποστηριχθούν, ε, οι αγώνες τους για την προστασία του δάσους του Αμαζονίου και την προστασία των δικαιωμάτων των ηθαγενών που ζουν στην περιοχή. Αυτοί οι απίστευτοι άνθρωποι θα πρέπει να ακουστούν. Οι άνθρωποι αυτοί χρειάζονται την άμεση υποστήριξή σας. Και τέλος, ενώ δεν ξέρω που βρίσκεται ο πατέρας μου, να πω ότι πιστεύω ότι είναι ζωντανός. Πιστεύω ότι το πνεύμα του όπως αποθανατίζεται από το βραβείο Ζαχάροβ τιμά τον πατέρα που ξέρω που έφερνε τον υπολογιστή του στην κρεβατοκάμερά μου όταν το χρειαζόμουν. Τώρα σας χρειάζεται ο λαός των Ουιγούρων. Σας ευχαριστώ. Thank you. Άρχεται η συνεδρία. Ο κύριο Τζαμπάσκι έχει δει το λόγο. Κύριε Πρόεδρε, ζήτησα το λόγο όπως το έκανε χθες και ο κύριος Φιλίπ Λατέρ και ο συνάδελφος Ερτούκ Μερικοί αισθάνθηκαν ότι προσευλήθησαν. Εντάξει, δεν υπάρχει πρόβλημα, ζητώ συγγνώμη. Εγώ ζητώ συγγνώμη, είμαι Βούλγαρος, ε, έχω ρίζες στη Σερβία, ακόμα και στην Τουρκία και δεν αν αισθάνονται οι δύο συνάδελφοι ότι προσευλήθησαν, τους ζητώ συγγνώμη. Αλλά δεν υπάρχει καμία συγγνώμη για τον τρόπο με τον οποίο δημιουργείται αυτό το πακέτο της πολιτικής για το περιβάλλον, της ε, ρήπανσης της ατμόσφαιρας ε, και για την πολιτική που δεν δημιουργεί ε, θέσεις απασχόλησης. Και ο τρόπος με τον οποίο οι Ευρωπαίοι αναθέτουν δουλειές στην Τουρκία και στη Ρωσία και γι' αυτό οι ίδιοι θα πρέπει κάποια να ζητήσουν συγγνώμη. Ευχαριστώ πολύ. Περνάμε λοιπόν στο δεύτερο γύρο εκλογής ε, του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή, του ή της Ευρωπαίου ή Ευρωπαίας Διαμεσολαβητή, κυρία Ντάλη. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Απλώς ε, να διορθώσω κάτι. Έχετε δικαίωμα να διαφωνείτε με το πακέτο για την κινητικότητα, το οποίο ε, δεν είναι η δική σας προσωπική άποψη. Αλλά σε καμία περίπτωση, ως Πρόεδρος τη Επιτροπής Μεταφορών αυτού του Κοινοβουλίου, με τον συνάδελφο Ισμαήλ Ερτούκ, δεν πρόκειται να ανεχτούμε τα όσα είπατε για, ε, για την καταγωγή μας, και την καταγωγή μου. Πρώτον, γιατί εσείς αποστέλλετε ένα ρατσιστικό μήνυμα και δεύτερον, ποτέ δεν πρόκειται να υποκύψω, θα μείνω όρθια, ούτω ώστε τέτοιε ε, ρήσει ποτέ να μην γίνονται δεκτέ σε αυτό το κοινοβούλιο. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε την πρόεδρο τη επιτροπή Μεταφορών, την κυρία Ντάλη. Και τώρα περνάμε στην, ε, στον δεύτερο γύρο εκλογής Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή. Σύμφωνα με το άρθρο 231 του κανονισμού θα κάνουμε τώρα ε, μια δοκιμή. Βέβαια είναι γεμάτη αίθουσα. Παρ' όλα αυτά πρέπει να κάνουμε αυτή τη δοκιμή γιατί έτσι προβλέπεται στον κανονισμό. Ε, να δούμε πώς είναι παρόντες γιατί χρειαζόμαστε ενισχυμένη παρουσία των Ευρωβουλευτών και θα ήθελα να ανακοινώσω ότι Νίλ Μούσνιετς έτσι ε, υποψηφιότητα του αποσύρθηκε. Έχουμε λοιπόν του εξή υποψήφιους Τζουζέπε Φορτουνάτο, Τζούλια Λαφράγκα, Έμιλι Οράιλι και Σεσίλια Βικ Κάνουμε λοιπόν τώρα τη δοκιμή. Άρχεται η συνεδρίαση. Η ψηφοφορία, με συγχωρείτε. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίζεται. Έκλεισε η ψηφοφορία. και βεβαίως έχουμε ε, την ικανοποιητική παρουσία των ευρωβουλευτών, την απαραίτητη παρουσία ευρωβουλευτών για να διεξαχθεί η εκλογή. Και θα ήθελα να επενθυμίσω ότι η ψηφορία είναι μυστική ε, και με βάση το 231 παράγραφος 6 του κανισμού ε, για να εκλεγεί ο υποψήφιος πρέπει να υπάρχει απαραίτητη πλειοψηφία. Οι αποχές δεν θεωρούνται έγκυρη ψήφος και από τη στιγμή που έχουμε τον κανονισμό 231 ε, 7 πριν ε, προχωρήσουμε στην εκλογή έπρεπε να γίνει δοκιμή έγινε η δοκιμή και έχουμε πράγματι τουλάχιστον 374 βουλευτές παρόντες έκλεισε η δοκιμαστική ψηφοφορία έχουμε όπως είπαμε τον, επαρκή, τον ικανοποιητικό αριθμό ευρωβουλευτών και η ψηφορία ε, θα γίνει ηλεκτρονικά. Σας έχουν δοθεί οι κάρτες, η ίδια διαδικασία όπως και χτες. Ε, θα βάλετε το όνομα του υποψηφίου και θα εκφράσετε την προτίμησή σας πατώντας το κουμπί μία και μόνο φορά. Είμαστε λοιπόν έτοιμοι. Ψηφίζουμε παρακαλώ. Ψηφίσατε όλοι. Έκλεισε η ψηφοφορία. Λοιπόν, ψήφισαν 694. Αποχές 56. 638 ψήφοι που κρίνονται έγκυροι, η απόλυτη πλειοψηφία 320. Ο Ράιλι 291. Λαφράγκ. 251, Φορτουνάντο 58, Βίξτρομ 38. Ως εκ τούτου ε, κανείς δεν ε, μπόρεσε να αποκτήσει τον, ε, την απαραίτητη πλειοψηφία για να εκλεγεί. Ως εκ τούτου, εφόσον κανένας υποψήφιος δεν έχει συγκεντρώσει την απαραίτητη πλειοψηφία, περνάμε τώρα στον τρίτο γύρο ψηφοφορίας ανάμεσα στους δύο πρώτους που είναι η κυρία Οράιλι και η κυρία Λαφράνκ. Ας αφήσουμε λίγο χρόνο για να μπουν τα ονόματα στους υπολογιστές μας. Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι. Ψηφίζουμε για Λαφράνκ και Οράιλι. Ψηφίζουμε παρακαλώ. La votazione è chiusa. Έκλεισε η ψηφοφορία. Λοιπόν, 694, 694 ευρωβουλευτές ε, έχουν δικαίωμα ψήφου, 94 αποχές, 600 ε, ψήφισαν, οι οράλοι 320 και οι οράλοι 280. Quindi sulla base del terzo turno di votazione proclamo ως εκ τούτου, με βάση τον τρίτο γύρο εκλογής, εξελέγει η κυρία Έμιλι Οράιλι και θα ήθελα να τη συγχαρώ, την κυρία Οράιλι. Θα προχωρήσουμε λοιπόν και στην επιβεβαίωση από πλευρά Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την εκλογή του Ευρωπαίου ε, Μεσολαβητή. Ο Επίτροπος κ. Χόγκαν έχει δει το λόγο. Uh, Κύριε Πρόεδρε, αγαπητή κυρία Οράιλη, θα ήθελα να σας συγχαρώ θερμά για την εκλογή σας σήμερα. Είναι πολύ εντυπωσιακή ένδειξη εμπιστοσύνης ε, από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και αναγνώριση του εξαιρετικού σας έργου τα τελευταία χρόνια ο θεσμός του Ευρωπαίου Διαμεσολευητή έχει γίνει πολύ σημαντικό ε, μέσο υλοποίηση των ευρωπαϊκών πολιτικών από την ίδρυσή του. Αποδεικνύεται ο ρόλος και η σημασία αυτού του ρόλου και χρήζει της αμέριστης στήριξή μας. Στα τελευταία χρόνια εμεί έχουμε ε, συμβάλει όσο μπορούμε στο να καταστήσουμε την ευρωπαϊκή διακυβέρνηση όσο γίνεται καλύτερη και πιο αποτελεσματική. Μόλις 5% των υποθέσεων ε, τελικά προκύπτει ότι υπάρχει κακοδιαχείριση και σε πάνω από 70% των ε, υποθέσεων η Επιτροπή ακολουθεί τι συστάσει του διαμεσολαβητή. Αυτό δείχνει ότι υπάρχει κλίμα εμπιστοσύνη και συνεργασία ε, μεταξύ των δύο θεσμικών οργάνων και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα συνεχίσει να είναι εταίρο που θα ενεργεί επικοδομητικά και θα ακολουθεί τι συστάσει, ε, λύσει και προτάσει σε ένα πνεύμα τέτοιο συνεργασία. Με έναν κοινό στόχο να βρίσκουμε τι κατάλληλε λύσει για του πολίτε μα. Ο Ευρωπαίος Δημοσιολαβητής και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχουν ένα κοινό συμφέρον να περνούν το μήνυμα ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα θεσμικά όργανα νοιάζονται για τους Ευρωπαίους πολίτες και τα προβλήματά, πολίτες τα προβλήματά τους. Κύριε Ωράιλη, και πάλι σα εύχομαι καλή επιτυχία στη νέα σα θητεία και η Επιτροπή και εγώ προσωπικά προβλέπουμε στη συνέχεια τη συνεργασία μα στο μέλλον. Ε, Ευχαριστώ τον Επίτροπο φυσικά να ευχηθώ καλή δουλειά στην Ευρωπαία Διαμεσολαβητή. Συνεχίζεται λοιπόν η ψηφοφορία. Και περνάμε στην ε, απόφαση για την ε, δημοσιονομική πειθαρχία από το 2021 και στην ε, ευελιξία όσον αφορά τους αριθμούς για το 2020 έκθεση Λίντς η προφορική ονομαστική ψηφορία άρχεται. Άρχεται η ονομαστική ψηφοφορία. Έκλειση ψηφοφορία. Εγκρίνεται. Ω εκ τούτου, ολοκληρώθηκε η πρώτη ανάγνωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Πάμε στην έκθεση ε, Κάρμεν Άβραμ. Πρόκειται για τη Συμφωνία Σύμπραξη Βιώσιμη Αλία Ευρωπαϊκή Ένωση Γκάμπια ε, και το πρωτόκολλο εφαρμογή τη. Έχουμε εδώ μία ονομαστική ψηφοφορία. Ψηφίζουμε παρακαλώ. Έκλεισε η ψηφοφορία. Εγκρίνεται. Περνάμε στην αντίρρηση, σύμφωνα με το άρθρο 112 του κανονισμού, είναι ονομαστική ψηφοφορία. Ψηφίζουμε παρακαλώ. Έκλεισε η ψηφοφορία. Εγκρίνεται. Περνάμε στο κλείσιμο των λογαριασμών ε, της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Υποστήριξης για το Άσολο για το οικονομικό του 2017. Υπέρ παρακαλώ ε, να σηκώσει το χέρι. Όποιος συμφωνεί, κατά, αποχές, οι λογαριασμοί έκλεισαν. Γίνεται ε, δεκτό αυτό, αυτή η έκθεση. Περνάμε τώρα στην έκθεση από πέντε πολιτικές ομάδες για τους ΛΟΑΔΜ. Πρόκειται για δημόσιες διακρίσεις και ρητορική μίσους κατά των ατόμων ΛΟΑΔΜ συμπεριλαμβανομένης της έννοιας των ζωνών χωρίς ΛΟΑΔΜ. Παράγραφος 3. Ονομαστική ψηφορία. Ψηφίζουμε παρακαλώ. Έκλειση ψηφοφορία. Εγκρίνεται. Παράγραφος 4. Χωρίστε σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα. Υπέρ παρακαλώ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται δεύτερο τμήμα, ονομαστική ψηφοφορία. Ψηφίζουμε. Έκλειση ψηφοφορία. Εγκρίνεται. Παράγραφος 6. Τροπολογία 11. Ονομαστική ψηφοφορία. Ψηφίζουμε παρακαλώ. Έκλειση ψηφοφορία. Εγκρίνεται. Παράγραφος 8. Τροπολογία υπεριθμών 2. Ονομαστική ψηφοφορία. Ψηφίζουμε. Έκλειση ψηφοφορία. Εγκρίνεται. Παράγραφος 12, ε, τροπολογία 3, ονομαστική ψηφοφορία παρακαλώ. Ψηφίζουμε. Έκλεισε η ψηφοφορία. <clears throat> Εγκρίνεται. Πάμε στην ε, παράγραφο 12, τροπολογία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 Έκλεισε η ψηφοφορία. Εγκρίνεται. Μετά την παράγραφο 23, τροπολογία 12, ονομαστική ψηφοφορία, ψηφίζουμε παρακαλώ. Έκλεισε η ψηφοφορία. Εγκρίνεται. Περνάμε τώρα ε, το 5, τροπολογία 5, υπέρ παρακαλώ, κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία υπερθμών 6, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Παράθεση 16, αρχικό κείμενο, ονομαστική ψηφοφορία. Ψηφίζουμε παρακαλώ. Έκλεισε η ψηφοφορία. Εγκρίνεται. Πάμε τώρα στην τροπολογία υπαριθμών 9, ονομαστική ψηφοφορία. Έκλεισε η ψηφοφορία. Εγκρίνεται. Εκτιμώντας ε, D, υπέρ παρακαλώ, κατά αποχές εγκρίνεται. Εκτιμώντας εν, τροπολογία 1, ονομαστική ψηφοφορία, ψηφίζουμε παρακαλώ. Έκλειση ψηφοφορία. Εγκρίνεται. Περνάμε στην ε, τροπολογία υπερθμών 13 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Εκτιμώντας ε, ο, τροπολογία 10, ονομαστική ψηφοφορία, ψηφίζουμε παρακαλώ. Έκλειση ψηφοφορία. Εγκρίνεται. Περνάμε στην ε, τροπολογία 14. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται τροπολογία 7 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται και περνάμε τώρα στην τελική ψηφοφορία για το ψήφισμα στο σύνολό του, ονομαστική ψηφοφορία. Ψηφίζουμε παρακαλώ. Έκλειση ψηφοφορία. 463 υπέρ εγκρίνεται. Και διαδικαστικό. Κάποιος έχει ζητήσει το λόγο. Δεν περάσαμε την ε, ψηφοφορία με ονομαστική κλίση για το εκτιμώντας Β στο αρχικό κείμενο. Όχι, το κείμενο είχε εγκριθεί προηγουμένως, άρα αυτή η ψηφορία κατέπεσε. Πάμε τώρα ε, στην απόφαση για την δίκαιη φορολόγηση ε, σε μια ψηφιοποιημένη και παγκοσμιοποιημένη οικονομία BEPS 2.0. Και περνάμε στην ε, τροπολογία 1 Ονομαστική ψηφοφορία παρακαλώ. Ψηφίζουμε. Δεκτή η τροπολογία. Παράγραφος 4. Ονομαστική ψηφοφορία. Ψηφίζουμε παρακαλώ. Έκλεισε η ψηφοφορία. Δεκτή. Τροπολογία 11. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Παράγραφος 9. Πρώτο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. Παράγραφος, ε, μάλλον δεύτερο τμήμα ε, της ίδιας ε, τροπολογίας. Ψηφίζουμε παρακαλώ. Έκλειση ψηφοφορία. Δεκτή η τροπολογία. Πάμε στην τροπολογία 8. Υπέρ, κατά, αποχές, Απορρίπτεται. Παράγραφος 12, τροπολογία 5 5Δ, 5 D, ονομαστική ψηφορία, υπέρ παρακαλώ. Ψηφίζουμε. Έκλειση ψηφοφορία. Απορρίπτεται. Και περνάμε στην τροπολογία 12, ονομαστική ψηφοφορία. Ψηφίζουμε παρακαλώ. Έκλειση ψηφοφορία. Απορρίπτεται. 13. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Η εννέα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Παράγραφος 23. Αρχικό κείμενο. Ονομαστική ψηφοφορία. Υπέρ. Ψηφίζουμε. Ψηφίζουμε. Έκλειση ψηφοφορία. Δεκτή. Τροπολογία 2. Ψηφίζουμε. Έκλεισε ψηφοφορία. Απορρίπτεται. Τροπολογία 14. Ονομαστική ψηφοφορία. Ψηφίζουμε. Έκλεισε ψηφοφορία. Απορρίπτεται. Αρχικό κείμενο σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές ε, δεκτό. Δεύτερο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. Παράγραφος 34. Αρχικό κείμενο υπέρ, κατά, αποχές γκρίνεται. Τροπολογία 3, ε, τροπολογία 3 ονομαστική ψηφορία. Ψηφίζουμε παρακαλώ. Έκλειση ψηφοφορία. Δεκτή. Τροπολογία 6 ονομαστική ψηφοφορία. Ψηφίζουμε. Έκλειση ψηφοφορία. Απορρίπτεται. Αρχικό κείμενο. Ονομαστική ψηφοφορία ψηφίζουμε. Έκλειση ψηφοφορία. Δεκτή. Τροπολογία 7. Ονομαστική ψηφοφορία. Ψηφίζουμε. Έκλειση ψηφοφορία. Απορρίπτεται. Αρχικό κείμενο. Ονομαστική ψηφορία. Ψηφίζουμε. Έκλειση ψηφοφορία. Δεκτή. Παράγραφο 41. Ονομαστική ψηφορία. Ψηφίζουμε. Έκλεισε η ψηφοφορία. Δεκτή. Περνάμε τώρα στην τροπολογία 15, υπέρ παρακαλώ. Κατά, αποχές, δεκτή. Παράγραφος 42. Αρχικό κείμενο, πρώτο τμήμα. Ονομαστική ψηφορία, ψηφίζουμε. Έκλειση ψηφοφορία. Δεκτή. Δεύτερο τμήμα, ονομαστική ψηφοφορία. Έκλειση ψηφοφορία. Δεκτή. Παράγραφος 43, ονομαστική ψηφοφορία. Ψηφίζουμε. Έκλειση ψηφοφορία. δεκτή. Η τέσσερα ονομαστική ψηφοφορία έκλεισε απορρίπτεται. Η 16 υπέρ κατά αποχές ε, απορρίπτεται. Η δεκαεπτά υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Η 10 σε δύο τμήματα ε, ψηφίζουμε παρακαλώ πρώτο τμήμα. Έκλειση ψηφοφορία. Απορρίπτεται. Δεύτερο τμήμα. Ψηφίζουμε. Έκλειση ψηφοφορία. Απορρίπτεται. Αρχικό κείμενο, ονομαστική ψηφοφορία. Έκλεισε. Δεκτή και περνάμε τώρα στην τελική ψηφοφορία. Ε, ψηφίζουμε παρακαλώ. Έκλεισε ψηφοφορία. Δεκτό το ψήφισμα. Πάμε στο επόμενο κείμενο που αφορά το κράτος δικαίου στη Μάλτα μετά τις πρόσφατες αποκαλύψεις σχετικά με τη δολοφονία της Ντάφνε Γκαρουάνα Γκαλίτσια. Ψηφίζουμε λοιπόν. Έκλεισε ψηφοφορία για την παράγραφο 8 δεκτή παρα, η τροπολογία. Τροπολογία 1, υπέρ παρακαλώ, κατά, αποχές, δεκτή, εκτιμώντας β σε δύο τμήματα, πρώτο τμήμα, υπέρ, κατά, αποχές, δεκτή, δεύτερο τμήμα, υπέρ, κατά,